που με το αξίωμα του Ευρωβουλευτή δεν είναι σύμβατο. Συγχαίρω του κυρίου Παντάρ και Ντεζίρ για του διορισμού του. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού διαπιστώνεται η χειρία των εδρών του από την 7η ή και από την 9η Απριλίου 2014 και θα ενημερωθούν οι αρμόδιε εθνικέ αρχέ για τη χειρία των εδρών. Οι αρμόδιε εθνικέ αρχέ με ενημέρωσαν για την εκλογή τη κυρία Κάτριν Ζάξ που από την 7η Απριλίου 2014 θα αντικαταστήσει τον κύριο Παντάρ. Το, άρθρο, σύμφωνα το κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 7 για την άμεση εκλογή των Ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 4, την εκλογή της κυρίας Σάξα από την 7η Απριλίου 2014 την έλαβε υπόψη και καλωσορίζω τη νέα ή παλαιότερη συνάδελφο και υπενθυμίζω σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ευρωκοινοβουλίου του Κανονισμού κάθε μέλος συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στα, στις